αυτή την ιδιότητά του. Οι αρμόδιες ελληνικές αρχές έθεσαν αίτημα για την άρση τη ασυλία του Ευρωβουλευτού κ. Σπύρου Δανέλη. Σύμφωνα με το άρθρο 6, εδάφιο 2 του κανονισμού, αυτή, αυτό το αίτημα θα διαβιβαστεί στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων του Ευρωκοινοβουλίου. Η Νομική Επιτροπή, στη συνεδρίασή της ε, στις 17 ε, Δεκεμβρίου 2012, εξέτασε την ε, εντολή νέων μελών και ομόφωνα πρότεινε να θεωρηθούν έγκυρες αυτέ οι εντολέ. Αφορά την κυρία Γιουστίνα Βιτκαουσκάιτ από την 21η Νοεμβρίου Νοεμβρίου 2012 και την κυρία Μόνικα Παναγιώτοβα από την 6η Δεκεμβρίου